przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Beginning of the... Έναρξης της Συνόδου της Ολομέλειας. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 10 marca. Λοιπόν, είχε διακοπή στις 10 Μαρτίου του 2011 η Σύνοδος και συνεχίζεται σήμερα. Τα πρακτικά και το κείμενο για τη Σύνοδο της 10ης Μαρτίου του 2011 έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν τυχόν σχόλια. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, οπότε θεωρούνται τα πρακτικά ως ε, εγκεκριμένα. Λοιπόν, τώρα κάποια σχόλια στην αρχή της ε, συνεδριάσεώς μας θα ήθελα να καλωσορίσω τη Μαρία Ρωμάνα Ντεκάσπαρη, τη θηγατέρα του μεγάλου ηγέτου Αλτσίντε Ντεκάσπαρη, που ήταν ένας από τους ιδρυτές πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Δεύτερη πληροφορία που έχω να σας δώσω. Ανησυχητικά νέα λαμβάνουμε από γειτονικές χώρες Μπαχρέιν, Συρία και Ιεμένη. Σε όλες αυτές τις χώρες οι διαδηλώσεις κατεστάλησαν ε, και ήταν άνθρωποι αυτοί που διαδήλωναν για περισσότερη δημοκρατία και στρέφουν οι κυβερνήσεις τα όπλα κατά του λαού τους και οι κυβερνήσεις αυτές χάνουν κάθε ε, δημοκρατική νομιμότητα θα πρέπει να σταματήσει η βία και αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα πρέπει ε, να δικαστούν. Επόμενο θέμα προ ενημέρωσή σα. Αυτή την εβδομάδα η διεθνή κοινότητα γιορτάζει την εβδομάδα αλληλεγγύη με τις χώρες που πολεμούν τον ρατσισμό και την διάκριση με ε, βάση ε, τη φιλετική καταγωγή. Τελευταία πολλά έχουν γίνει στον ελεύθερο κόσμο για να εκριζωθεί ο ρατσισμός από την καθημερινή ζωή. Ξέρουμε ότι πολλά απομένουν πρέπει να γίνουν και στα κράτη-μέλη και εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άλλο ένα θέμα προς ενημέρωσή σας. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα μάθαμε ότι ένας από τους συναδέλφους μας, ο κύριος Τάλερ, παρετήθηκε από τη θέση του στο Κοινοβούλιο και δεύτερος συνάδελφος, ο κύριος Στράσερ, και εκείνος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη θέση του τις επόμενες μέρες. Τρίτο μέλος, ο κύριος Σεβερίν, αποχωρεί από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.